Συγχαίρω τον κύριο Κοφεράτη για την εισήγησή του. Ευχαριστώ κύριε Σβάμπ. Απλώς να επιβεβαιώσω, ναι, περιμέναμε να έχουμε ε, αυτή την υποστήριξη. Το είχαμε ε, υποσχεθεί για το τέλος του έτους. Ο Βάνος, ο επικεφαλής της μονάδας μου, είπε ότι υπήρξε αναβολή διότι δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από το πρώτο σχέδιο. Ελπίζω τον επόμενο μήνα να την έχουμε αυτήν την μελέτη και να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε και να την εντάξουμε στο τελικό πακέτο τροπολογιών για την εισήγηση του κυρίου Κοφεράτη. Θα συζητήσουμε και την ιδέα να παραγγείλουμε κάποια συμπληρωματική εργασία για τους μακροπρόθεσμους δείκτες απόδοσης και αντικτύπου της ενιαίας αγοράς. Ε, η κυρία Στάιλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σχετικά με τους δείκτες. Χαιρετίζουμε την ιδέα αυτή. Όταν αναφέρεται το θέμα ε, της αξιολόγησης αντικτύπου, εάν αυτοί οι δείκτες όταν αναπτυχθούν θα μπορούσαν να περιληφθούν στην αξιολόγηση αντικτύπου. Όταν εξετάζουμε τα, τις νομοθεσίες θα πρέπει να δούμε ε, ποια, ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών στην ενιαία αγορά. Βεβαίως αναφέρθηκαν οι θέσεις αγορά στην ενιαία αγορά Άλλοι μίλησαν για το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν ε, τα μέσα αυτά. Και σχετικά με τα προϊόντα οικοδομών είναι ένα σημαντικό ε, θέμα για τις κατασκευές και νομίζω ότι οι ετήσιες εκθέσεις που έχουμε είναι σημαντικές ε, επειδή επισημαίνουν θέματα όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά, ελλείψεις και βλέπουμε ότι εκεί όπου τα κράτη-μέλη εφαρμόσουν τους κανόνες της ενίας αγοράς υπάρχει αντίκτυπος και ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη για την εισήγησή του και άλλους που συνέβαλαν και χαίρομαι ε, που είχαμε το θέμα αυτό σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχω μια κάπως διαφορετική άποψη, διότι είναι τα Χριστούγεννα και τα δέντρα των Χριστουγέννων περιλαμβάνουν τα πάντα. Κρέμονται πάρα πολλά στολίδια και αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο προσπαθεί να συντονίσει τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε στην πραγματική οικονομία. Αν βάλουμε πολλά πράγματα, δεν θα έχουμε αρκετά στο τέλος. Ελπίζω ότι έχετε επαφές με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι τόσο ευτυχής σχετικά με αυτές τις συστάσεις ε, και ό,τι έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς, ε, η χώρα μου δεν είναι στην Ευρωζώνη, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτές τις συστάσεις αλλά 17 ή 18 χώρες είναι στην Ευρωζώνη και θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις, αλλά δεν το πράττουν. Αυτό είναι ίσως ένα άλλο πρόβλημα. Αυτό είναι από αυτό που λέω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ε, ε, πλησιάζουμε το θέμα της, ε, της κυριαρχίας. Πολλοί από εμά υπήρξαμε μέλη εθνικών κοινοβουλίων ε, και αυτόμεθα της εθνικής κυριαρχίας πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε τα πάντα, να λέμε κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, η πιο γενική παρατήρηση. Και η δεύτερη είναι το άρθρο 16 εδώ που αναφέρεται στην κινητικότητα, στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί και να σας ζητήσω από εσά κύριε Πρόεδρε να, να διαβιβάστε κάποιο μήνυμα στο Λονδίνο. Ήμουν στο Λονδίνο πριν μερικές εβδομάδες προτού διαβάσω το άρθρο του κυρίου Κάμερον και άκουσα την ομιλία του φιλελεύθερου ηγέτη επίσης και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι επικίνδυνο. Έχουμε την ίδια ρητορική σε πολλές χώρες μας και αυτό δεν βοηθά καθόλου την ενιαία αγορά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω είναι ότι αυτοί οι δείκτες ισχύουν για όλες τις χώρες, όχι μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης. Και το θέμα μας για το εξάμεινο είναι το γεγονός ότι για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να αυξήσουμε τις οικονομικές επιδόσεις θα πρέπει να αποδίδουν καλύτερα οι οικονομίες μας, όπως είπε η κυρία Στάιλερ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι για την ώρα θα πρέπει να εστιαστούμε στους οικονομικούς δείκτες ε, και να δούμε επίσης και την ε, επίδοση της ενιαίας αγοράς. Όταν πήγαμε στην Ελλάδα, όσοι πήγαμε αποστολή στην ε, Ελλάδα, είδαμε ότι με αυτό το θέμα ασχολείται τώρα η ελληνική κυβέρνηση, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός και επίσης αυτό δεν ήταν μόνο ένα θέμα διεξιάς αριστεράς, διότι όταν είδαμε τις ε, συνδικαλιστές στην Ελλάδα λένε το ίδιο πράγμα. Έχουν πλήρη συνείδηση αυτού του γεγονότος. Οι οργανώσεις καταναλωτών επίσης έχουν συνειδητοποιήσει ε, το θέμα ότι δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός και οι καταναλωτές έχουν λιγότερη επιλογή. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε, αλλά συμφωνώ μαζί σας, αν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσματική οικονομία θα πρέπει να έχουμε περισσότερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Μήπως υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο σχετικά με την εισήγηση του κυρίου Κοφεράτη ενώ έχετε τη δυνατότητα. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας ενημερώσω για την δυνατότητα να υπάρχει έκθεση για αυτό το θέμα. Εγώ προσωπικά χαιρετίζω μια τέτοιου είδους μελέτη, αλλά ήδη επισήμως έφτασε πάρα πολύ αργά αυτό το αίτημα. Προβλέπουμε για, την, για όλο το χρόνο 10 με 10, με 10 με 12 τέτοιου είδου σχέδια. Πήραμε αποφάσεις για 6 έρχεται αυτή η θητεία Πρέπει να θα δώσουμε στους επόμενους συναδέλφους. Εάν ήδη το απεφάσισε για τα έξι, το θέμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές δυνατότητες για μια τέτοια μελέτη. Πρώτα απ' όλα να τη χρηματοδοτήσουμε τους ιδίους πόρους της Επιτροπής μας και δεύτερον μέσω της διεύθυνσης έρευνας του Κοινοβουλίου που κάνει μελέτες αξιολόγησης. Άρα, εφόσον το χρειαζόμαστε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μία καλή μελέτη, ούτως ή άλλως, που θα μας χρησιμεύσει και πέραν της έκθεσης Κοφεράτη. Κύριε καθηγητά Κορέα Κέμπος, Σε επαφή με τον Διευθυντή της ε, Διεύθυνσης ε, Έρευνας Τεχνολογίας και θα δούμε κατά πόσον θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την μελέτη για τους δείκτες και την καινοτομία που είναι τόσο σημαντική. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε τα πράγματα να τα δυσκολεύσουμε. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό μεταξύ των συντονιστών για να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ καλύτερους δείκτες επιδόσεων για την ενιαία εσωτερική αγορά από αυτούς που διαθέτουμε τώρα. Κυρίως να δούμε πώς έχει μεταφερθεί ε, ε, ε, έχουν μεταδειχθεί κοινοτικέ οδηγίε στην εθνική αγορά και να δούμε κατά πόσον υπάρχουν ελλείψεις. Και νομίζω ότι τέτοιου είδου δείκτες δεν τους χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά για να δούμε πώς λειτουργεί τελικά η αγορά για τους καταναλωτές. Επίσης και η μονάδα στατιστικών ε, ενδιαφέρεται τη μετάσχη. Πράγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συντονιστούμε. Θέλει κανείς σας το λόγο. Σε αυτή την περίπτωση θα δώσω και πάλι τον λόγο στον εισηγητή κύριο Κοφεράτη να ολοκληρώσει και μας υπενθυμίσει προθεσμίες κατάστασης τροπολογιών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις διευκρινήσεις και τα σχόλια. Τόσο τους Σκιώδης, όσο και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Επειδή το κλίμα είναι χριστουγεννιάτικο, δεν θέλω να υπάρξουν πρόσθετες ανησυχίες. Κυρίως για τον κύριο Όλη και το χριστουγεννιάτικο δέντρο του. Υπάρχει μια μεσογειακή, ένα μεσογειακό έθιμο που συνήθως ε, συνίσταται στο να στολίζουμε φάτνη τα Χριστούγεννα. Μια φάτνη που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό είναι πολλαπλά τα επιχειρήματα. Προκειμένου όμως να αποφύγουμε τάχη, δεν θα σχολιάσω όλες τις παρατηρήσεις, απλώς δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, συμμερίζομαι απολύτως την ανάγκη να συμπληρωθεί άμεσα η μελέτη η οποία παραγγέλθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έκθεσης ΣΒΑΜ γιατί όντως χρειαζόμαστε δείκτες, δείκτες που σήμερα να μας επιτρέψουν ίσως όχι για την έκθεση αυτή γιατί δεν προλαβαίνουμε αλλά τέλος πάντων για τα επόμενα βήματα ένα τρόπο να μετρούμε τα στοιχεία της εσωτερικής, της ενιαίας αγοράς και να βλέπουμε ποια είναι τα ωφέλη ή που υπάρχουν περιορισμοί βάσει γνώσεων, στοιχείων που δεν θα είναι μόνο ποσοτικά αλλά να βλέπουμε και την αποτελεσματικότητα των δράσεων και την ποιότητά τους δηλαδή. Σήμερα διαθέτουμε, δεν διαθέτουμε ακόμα μέσα οι εργαλεία, οι δείκτες που έχουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Το λέω για όσους θα μας διαδεχτούν ή για όσους θα παραμείνουν στην επόμενη θητεία το μέλλον της εσωτερικής αγοράς δεν αποτελείται μόνο από συστάσεις ή από πολιτικές εντολές αλλά και από δράσεις πολύ χειροπιαστές. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε στους υπόλοιπους τη σημασία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της εσωτερικής αγοράς. Και αυτή η συζήτηση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο αντιμετωπίζει αντιστάσεις και από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και από την Επιτροπή Απασχόλησης ακριβώς για τον λόγο αυτό. Διότι ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί ποια είναι η αξία και η σημασία των δράσεων που αποφασίζει η Επιτροπή μας είναι πιο απλό. Ας κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να συμμετάσχουμε στις δράσεις και τους στόχους και οι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται, αλλά θα πρέπει εμείς να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες τους και να ενδυναμώσουμε αυτές τις δράσεις. Η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά είναι η δική μας εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με την εσωτερική αγορά και δράση με τη δράση, τομέα με τον τομέα, πρέπει να δείξουμε ποιο είναι το ποιοτικό άλμα που έχει γίνει με την υλοποίηση των πολιτικών της εσωτερικής αγοράς. Δεύτερη παρατήρηση, η οποία είναι σχετική με την προηγούμενη. Αντιλαμβάνομαι απολύτως και γι' αυτό ζήτησα κάποιες ε, διευκρινήσεις για ποιο λόγο Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων, το θέμα αυτό το καλύψαμε ήδη. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά κατά την άποψή μου η Επιτροπή μα έχει οριζόντιε αρμοδιότητε. Δεν μπορεί να ασχολείται με συγκεκριμένα περιορισμένα θέματα, σίγουρα και με κάποια περιορισμένα θέματα, αλλά αναπόφευκτα πρέπει να καλύψει και θέματα άλλων επιτροπών που είναι αρμοδιότητα άλλων επιτροπών. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, ε, όποια υπέρβαση των ορίων υπάρξει, χρήσιμη θα είναι. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε από τα χέρια των άλλων τη δουλειά του. Απλώ βρίσκουμε του συνδετικού κρίκου μεταξύ αυτών που κάνουν οι άλλοι και αυτών που κάνουμε εμεί. Και εκείνοι που με ζήλο επερασπίζονται τα σύνορα των αρμοδιοτήτων τους δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε διότι θα μπορούσαμε ε, με ε, απόλυτη ε, ευθύνη να κάνουμε κάποια τέτοια υπέρβαση των ε, ορίων αυτών των εντό εισαγωγικών συνόρων και να προσφέρουμε πολλά όπως έγινε με, την ευρωπαϊκή, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο διότι οι άλλοι μπορεί όντως να μην προωθήσουν αρκετά την εσωτερική αγορά στο το κάναμε εμείς. Μην ξεχνάμε ότι για τα εθνικά κοινοβούλια είναι πιο σημαντικό αυτό που βασίζεται εδώ αυτό που από αυτό που αποφασίζεται σε άλλες επιτροπές. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά αυτή είναι η πρόσθετη αξία της επιτροπής μας. Και τελικά δεν αναγνωρίζεται το έργο μας. Γι' αυτό λοιπόν επέτρεψα στον εαυτό μου να γράψω κάποια πράγματα που ίσως ξεπερνούν ελαφρώς τα όρια των αρμοδιοτήτων μας. Πάντως η αρχική πρόθεση ήταν αυτή. Και μετά συζητούμε από κοινού αν πρέπει ή όχι να προχωρήσουμε. Αλλά μην παραμείνουμε αποκλεισμένοι σε ένα τομέα όπου ένα μέρος της δουλειάς μας εν τέλει δεν δίνει τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να αποκομιστούν. Σε ό,τι το πώς θα συνεχιστεί πορεία της εκθέσης αυτής και ας με διορθώσει ο Πρόεδρος, εάν κάνω κάπου λάθος, θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 23 Ιανουαρίου, μετά να πάμε στην Ολομέλεια, στα μέσα Φεβρουαρίου, οπότε ο χρόνος που έχουμε δεν είναι πολύς, όμως η κατάσταση και η πρόοδος της με όσα είδαμε να γίνονται με την έκθεση Σβάμπ, αλλά όσα γίνονται και τώρα πιστεύω ότι είναι αντικείμενο συμφωνίας από όλους ιδίως γιατί μπορούμε να συμπληρώσουμε και το έργο άλλων επιτροπών. Ευχαριστώ. that's exactly correct. Um, Πολύ σωστά. Στις 9 Ιανουαρίου όταν θα επανέλθουμε μετά από τις ε, χριστουγεννιάτικες διακοπές θα στήσουμε τις ε, συμβεστικές τροπολογίες και για την έκθεσή μας μαζί με την έκθεση των, ε, της Επιτροπής της Απασχόλησης προβλέπεται να συζητηθεί το θέμα αυτό στην δεύτερη ονομέλεια του Φεβρουαρίου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλοι να συμμετάσχουμε τώρα. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας πριν αρχίσουμε την ε, ψηφοφορία. Σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν στο τέλος του 2013 να κάνουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Ο φωτογράφος είναι εδώ. Παρακαλώ λοιπόν όλα τα μέλη καθώς και τους αναπληρωτές, τακτικά μέλη και αναπληρωτές, να έρθουν εδώ στη μέση της αίθουσα για να κάνουμε την ε, οικογενειακή φωτογραφία για να στολίσετε μαζί με τις άλλες χριστουγεννιάτικες κάρτες που θα έχετε. Okay, um, let's make a start. Ας αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο Ροσφόρ, με την έκθεση του κυρίου Ροσφόρ για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και την σχετική οδηγία. Θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς και μόνον, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι μετά από την συζήτηση τη χθεσινή, ε, παρά το γεγονός ότι είμαστε σύμφωνοι, συνεχίζουμε τις συζητήσεις μέχρι αργά το βράδυ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γι' αυτό. Πολύ καλά. Άρα υπάρχει περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα των συμβιβαστικών προτάσεων. Θα κάνουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιος είναι ο υπεύθυνος ε, των σοσιαλιστών? Εσείς. Οκ. Okay. Λοιπόν, να μου το λέτε. Λοιπόν, ε, τροπολογία 1 για να 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. 30 ψήφισαν. Έρχεται και ο κύριος Αρίας. 31 συνάδελφοι ψηφίζουν. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 15 προς 15.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 Εγκρίνεται, αλλά δεν είναι απολύτως σαφές. Κύριος Μάιερ, 15 προς 16, απορρίπτεται, 8, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε στην ε, τροπολογία 1 της ε, Τζούρι. Επιτροπή Ζωμικών Υποθέσεων. Αρχίζει η ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 14 και 18, αποσύρεται οι 25, φτάνουμε στην 17, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 19 καταπίπτει, 24 καταπίπτει, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα στην τζούρι 5. Τζούρι 5 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 3 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά αν θέλετε κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ας το κάνουμε λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τζούρι 4 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Καταπίπτει. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 6. Υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω όμως ότι εγκρίνεται. Λίγη ψηφοφορία. 17 προς 13 εγκρίνεται. 14 με τον κύριο Μάγερ. 7 της Τζούρι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τζούρι 8 προστίκη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 5, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τζούρι 9 ως προσθήκη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7, χωριστή ψηφοφορία που έχει ζητήσει η ECR. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος, δηλαδή χωρίς την ε, τελευταία πρόταση, έτσι όπως αναφέρεται και στο εγγραφό σας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56. Καταπίπτει. 47. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, ε, ε, όχι, όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη, 55, ψηφίζουμε την 55. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 της κυρίας Ενάλοβα, χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 60. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Τώρα αρχίζει η ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης έτσι όπως την τροποποίησαμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία και εγκρίνεται με 32 ψήφους. Ομόφωνα. Ευχαριστούμε κύριε Ροσφόρ. Ελπίζω ότι στην Ολομέλεια θα έχουμε μια πολύ παρουσίαση του θέματός μας για να είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε έγκριση εκθεσής μας. Φτάνουμε τώρα στην επόμενη εκθέση της κυρίας Κόλιν Λάγκεν. Νομοθετική πρόταση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Θέλετε να λάβετε το λόγο κύριε Κόλιν Λάγκεν. Ναι κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω να ψηφίσουμε την εντολή για να μπορέσουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να κερδίσουμε χρόνο. Διότι πριν από το τέλος Ιανουαρίου, όπως ξέρετε, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για να περάσουμε στα επόμενα στάδια. Μετάφρες και όλα αυτά. Πολύ καλά. Εάν ε, ψηφίσουμε πρώτα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ψηφοφορία και αν συμφωνήσουν μετά οι συντονιστές, όντως θα σας δώσουμε με τον κλασικό, σωστό τρόπο την ε, εντολή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κύριε Σφάπ, κύριε Κρότζερ, κύριε Σαντομόζερ, βλέπω ότι συμφωνείστε. Κυρία Ρούλε επίσης συμφωνεί. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν. Λοιπόν, ας περιμένουμε την ε, τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Άρθρο 1, Τροπολογία 54 υπέρ κατά απορρίπτεται. 55 προφορική υπέρ κατά επαναλαμβάνω υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 είναι προσθήκη στο 56, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 αποσύρεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 αποσύρεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 ως προσθήκη. Υπέρ. Ε, θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 66. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 69. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 16 προς 16, 73 του κύριου Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, 5, τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 3 του εισηγητή, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 όχι, συγγνώμη, 9 του εισηγητού, όλες οι άλλες καταπίπτουν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 του κυρίου Κρόιτσμαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, Υπέρ. Υπέρ του 45. Κατά. Εγκρίνεται. 46. Αποσύρεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 της εισηγήτριας και της κυρίας Ρούλε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51, υπέρ, υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την, ε, το σχέδιο έκθεσης έτσι όπως το τροποποίησαμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα σχεδόν με μόνο μία ψήφο κατά συγχαρητήρια. Λοιπόν, σύμφωνα με το έντιμα της κυρία Κόλιν Λάγκε και επειδή συμφωνούν οι συντονιστέν, θα ήθελα να μας αναθέσετε την εντολή να διαπραγματευτούμε με την Προεδρία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αρχίζει η ψηφοφορία και για να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εντολή θα πρέπει να έχουμε 21 ε, συν 1 ψήφους. Ω, 31, 31. Τέλεια. Τέλεια. Σαφέστατη εντολή. Καλή τύχη στην πρώτη σας νομοθετική έκθεση. Και όπως πάντα θα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε τακτά διαστήματα και σε όλες τις συνεδριάσεις μας. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Επιτροπής του Συμβουλίου. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι. Όχι. Είναι παρόν και το Συμβούλιο. Η Προεδρία. Η επόμενη, η επόμενη Προεδρία είναι εδώ. Η επόμενη Προεδρία είναι παρούσα. Χαιρετίστε μας να σας δούμε. Λοιπόν, σας ε, καλωσορίζουμε θερμά και θα σας δούμε περισσότερο το επόμενο εξάμεινο και χαιρετίζουμε τη συνεργασία μαζί σας. Πολύ καλά. Η επόμενη έκθεση. Η έκθεση του κυρίου Αρίας πρόταση πρωτοβουλία για ολοκληρωμένη αγορά παράδοση δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να πει κάτι ο εισηγητή, Όχι. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. We start with compromise amendment 1. Those in favour, those against, abstentions, that's carried. Uh, amendment 9 as an addition, those in favour, Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, μεταφορές 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. με εγκρίνεται 17 προς 15. 10... Μεταφορές 5, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, μεταφορές 2, τρανς 2, υπέρ κατά ε, εγκρίνεται, συμβαστική 9, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 14 καταπίπτει. 29 καταπίπτει. την Επιτροπή Απασχόλησης, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος να ελέγξουμε εδώ ότι ψηφίζουμε σωστά. Συμβιβαστική 6. για την 32 θέλω κάτι να πω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 Compromise Amendment 5. So we're now we're on, on Compromise Amendment 6. Those in favour? Those against? Abstentions? That's carried. So I'm now on Amendment 43. Those in favour? Αποχές απορρίπτεται. 44. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 46 εγκρίνεται, τραν 11, υπέρ κατά απορρίπτεται, 48 υπέρ κατά εγκρίνεται, 49 αποσύρεται, συμβιβαστική 7, προφορική τροπολογία ο κύριος Αρίας θέλει κάτι να πει. Για την προφορική τροπολογία στην συμβιβαστική 7 δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να την εγκρίνω δεδομένου ότι ήδη με όλες τις ομάδες είχαμε καταλήξει σε συμβιβασμό και σε αυτή την περίπτωση δεν συμφωνούμε όλοι με τη συμπερίληψη. Για να μην χαλάσει λοιπόν ο συμβιβασμός τον οποίο είχαμε καταλήξει είμαι αντίθετος σε αυτή την προφορική τροπολογία, άρα θα πρότεινα να μην τη συμπεριλάβουμε στην ψηφοφορία. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε γιατί περισσότερο από δύο μέλη δεν τη δέχονται, λέει ο πρόεδρο. Πολύ καλά. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβαστική 7 χωρίς την ε, προφορική αυτή τροπολογία. Χωρίς, χωρίς την προφορική. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τραν 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τραν 12. Όχι, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική 10. Το 9 τι έγινε, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 12. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται, 58 υπέρ κατά εγκρίνεται, 59 υπέρ κατά ε, ξαναψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται 60 υπέρ κατά εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη, ε, τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά απορρίπτεται, 5 υπέρ κατά εγκρίνεται, 6 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται, αποσύρεται η 7 Τροπολογία 1 υπέρ κατά απορρίπτεται και ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο έκθεσης έτσι όπως την τροποποίησαμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ομόφωνα εγκρίνεται με 33 ψήφους. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια. θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι τέλεια και η παρουσία στην Ολομέλεια. Περνούμε τώρα στην επόμενη έκθεση. On the um, directive on rules on pressure equipment, um, uh, this is really the Εναρμόνιση των νομοθεσιών των 100 μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υποπίεση. Έκθεση της κυρίας Ρόιτοβα. Να αφήσω την κυρία Ρόιτοβα να μας πει το ιστορικό της πρότασης και μετά ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες on block. Απλώς εξηγήστε μας που βρισκόμαστε σε σχέση με το όλο πακέτο. Κυρία Ρόιτοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνεργασία με όλους τους σχέδιους εισηγητές ήταν εξαιρετική και χάρη ε, στη συνεργασία της Προεδρίας μας μπορέσαμε να φτάσουμε στο, στην επίλυση του όλου θέματος. Το πακέτο αυτό που είναι ουσιαστικά η πολλωστή οδηγία για τα θέματα αυτά θα μας δίνει τη δυνατότητα να, τα, να υλοποιήσουμε τα προβλεπόμενα μέτρα. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ε, τροπολογίες, οι οριζόντιες αλλαγές είχαν ήδη εγκριθεί από άλλες οδηγίες. Οπότε οι τροπολογίες δεν επέφεραν επί της ουσίας τροποποίηση. Έκανα και εγώ αρχικά κάποιες προτάσεις που μου φαίνονταν εύστοχες, αλλά δεν επέμεινα. Ε, ε, έπειτα χρειάστηκαν κάποιες διευκρινήσεις, συγκεκριμένα μια γλωσσική διόρθωση και υπάρχουν και τρεις ε, ακόμη γλωσσικές τροπολογίες όπου απλώς προσαρμόζεται το κείμενο στη διατύπωσή του. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε πραγματικά on block συνολικά τις τροπολογίες. Το συζήτησα και με τους σκιώδεις εισηγητές και θα πάρω το λόγο στο τέλος της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος από τους κοιόδες να σχολιάσει. Βέλος προχωράμε στην ψηφοφορία. Ωραία. Όλες οι τοπολογίες μαζί. Ο μπλοκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Τελική Έκθε... ε, ψηφοφορία η κυρία Ρότοβα. Θέλετε τώρα το λόγο ή να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε δύο δεν ψηφίζουν δεν πειράζει πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται 30 υπέρ καμία ψήφος κατά Θέλατε το λόγο ναι, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο για μένα. Θα ήθελα λοιπόν να μου αναθέσετε και τη διαπραγματευτική εντολή για να μπορέσω να προχωρήσω σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Έλαβα επιστολή από το Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί όλη η προσπάθεια σε μια από τι επόμενε ολομέλειε. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ανάθεση μια διαπραγματευτική εντολή με το Συμβούλιο και ζητώ από τον Πρόεδρο να ψηφιστεί αυτή η διαπραγματευτική εντολή για να μπορέσουμε να έχουμε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ναι, να επιβεβαιώσω ότι οι σκιώδεις εισηγητές συμφωνούν με όλα αυτά, διότι ουσιαστικά θα συνεχίσουμε τη δουλειά που έχει ξεκινήσει. Ίσως να χρειαστεί και ένας μόνο διάλογος ε, για να ολοκληρωθεί αυτό. Εγώ συμφωνώ. Η ομάδα να παραμείνει η ίδια, αλλά ας γίνει επίσημη ψηφοφορία για να βεβαιωθούμε ότι όλοι συμφωνούν. Εντολή για την κυρία Ρόιτοβα λοιπόν. Πέρας. Είναι πολύ σαφέ. Έχετε την εντολή, κυρία Ρόιτοβα. Σα ευχαριστούμε πολύ και σα ευχόμαστε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην ε, τελική πρόταση του κυρίου Σμιτ. Ζητήσαμε χθε τι συμβαστικέ τροπολογίε. αποζημίωσης. Ο κύριος Φάμπ έχει αποσύρει κάποιες από τις τροπολογίες του, ενημερώνομαι. Οπότε έχουν αποσυρθεί αν είναι ακόμα στην, ε, στον κατάλογο των ε, τροπολογιών σας της ψηφοφορίας. Κύριε Σμίτ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, ωραία, οπότε προχωρούμε. 36 υπέρ κατά Αγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά Αγκρίνεται. συμβαστική 1 υπέρ κατά Αγκρίνεται. 42 υπέρ να ελέγξουμε 42 του εισηγητού. Πέρας. Εγκρίνεται 17 υπέρ 15 κατά. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 44 με συγχωρείτε. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 45 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47. Αποσύρθηκε. Αυτό σημαίνει όχι, ε, όλο το σύνολο αυτό το που πάμε, 48 ωραία, αποσύρθηκε όλο μαζί 48 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 50 αποσύρεται. 51 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 54 αποσύρεται. 55 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 56 και 57, 58 και 59 αποσύρθηκαν. 60 υπέρ. 60 υπέρ. Κατά. 61 αποσύρεται. 62, 63 και 65 της κυρίας Γράπτη unblock υπέρ κατά απορρίπτονται 64 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 αποσύρεται 66, 67, 68 καταπίπτουν 11 από τον εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. 69 υπέρ να ελέγξω. Απορρίπτεται νομίζω. Εξαρτάται αρκεί να ψηφίσουν όλοι. 32 ψήφισαν. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 70 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ίδια πλειοψηφία. 71 υπέρ κατά εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεν είναι σαφές. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία απορρίπτεται. 14 προς 18. 75. 75. Νομίζω να ψηφίσουμε και για αυτήν ε, ηλεκτρονικό. 75. Πέρας. Εγκρίνεται. 76 καταπίπτει. 77 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 80 ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Έλεγχο. Όχι, συμβαστική τρία. Συμβαστική τρία. Υπέρ. Να ψηφίσουμε, να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς γιατί είναι σημαντικό. Ε, συμβαστική τρία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 91 άρθρο 17, ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. 92. πέρασε. Έφυγαν τα αποτελέσματα από την οθόνη. Ψηφίστε ξανά παρακαλώ, συνεχίστε να ψηφίζετε. Πιέστε τα κουμπιά. Δεν ψήφισαν άπαντες. 31 κάρτες. 30 ψήφισαν. Εντάξει, πέρας Απορρίπτεται. Και 93 υπέρ. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογικέ σκέψει. 1 του συγκριτού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Έχει ήδη ψηφιστεί 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά εγκρίνεται. 17 καταπίπτει. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 και 22 εγκρίνονται. Αυτομάτως 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 23-24 εγκρίνεται μάτος 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 25 αυτόματο. 26 υπέρ κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 ψηφιστή 4 αποσύρεται 30 31 5 5 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 το εισηγητό υπέρ κατά εγκρίνεται 34 κατά πίπτη 7 υπέρ κατά Αγκρίνεται. 35 καταπίπτει. 8 τελευταία τροπολογία υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Σμιτ. Εντάξει, εγώ ήμουν η αποχή και δεν ψηφίστηκε η τροπολογία μου. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσει η συνάντηση των συντονιστών. Απλώς οι συντονιστές να μου πούν θέλετε να ξεκινήσουμε αμέσω, γιατί κανονικά ξεκινούμε στι 11 και 4. Αλλά νομίζω είναι όλοι εδώ, και ο κύριο Μάντερ, και ο κύριο Φαμπ, και η κυρία Σαλδεμόζε, η κυρία Ρούλε, και εγώ. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε την συνάντηση των συντονιστών στι 10 και 45 παρακαλώ, σε 5 λεπτά. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευχαριστώ πολύ για την δουλειά σα. Θα σα δω το Γενάρη.